presidente de Timor-Leste. Ο του Ανατολικού Τιμόρ. Welcome to the European Parliament. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε και πάλι, μετά από 18 χρόνια.